Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και στην Επιτροπή Ιστορική Αγορά η συζήτηση για την τομέα τη οικοδομή και εμεί θα τον παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ. Ευχαριστώ κυρία Στήλε. Απευθύνατε και προτάσεις στο Προεδρείο, τις οποίες σημειώσαμε. Η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να ε, το συζητήσει και να έχει μια απάντηση για το θέμα σας. Η συζήτηση έληξε εδώ. Ε, και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της στην ημερήσια διάταξη, που είναι δήλωση της Επιτροπής με θέμα «Συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εντοπισμό διοξίνης στι ζωοτροφές». Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Ντάλη. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το νέο έτος ξεκίνησε με ένα σοβαρό συμβάν. Είχαμε μόλυνση διοξίνης ε, ζωοτροφών στη Γερμανία. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, σε πλήρη μάλιστα συνεργασία με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Ήδη ξεκίνησα να σκέφτομαι τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να υπάρχει ένα σύστημα ε, ακόμη πιο αποτελεσματικό για ασφαλείς και υγιεινές ζωοτροφές. Ας ξεκινήσουμε όμως από το συμβάν. Το συμβάν ε, ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ενημερώθηκαν ε, στις 22 Δεκεμβρίου γερμανικές αρχές του, αφού έλαβαν τα αναλυτικά αποτελέσματα όταν ένα δείγμα συγκεκριμένα βρέθη να μην ε, συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μετά από δοκιμές αυτοελέγχου. Μετα, από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου πέρυσι. Ο κατασκευαστής έδωσε 7 αποστολές λιπαρών οξέων που προορίζονταν ε, για σε έναν μάλλον κατασκευαστή, ο οποίος επίσης παρασκευάζει ζωοτροφές. Μια εταιρεία η οποία ήταν και εγγεγραμμένη ως ε, παρασκευαστή ζωοτροφών. Μάλλον υπήρξε μια ανάμιξη από ό,τι φαίνεται ζωοτροφών με τεχνητές ε, ζωοτροφές και βρέθηκε στη συνέχεια ε, μόλυνση από δύο ξύνες. αλλά σε ελέγχους που κάναμε σε αρχές Δεκεμβρίου δεν βρήκαμε ε, άλλα κρούσματα. Πρέπει μέχρι όμως να υπάρξει επαλήθευση και για λόγους προληπτικούς όλες οι αποστολές αντιμετωπίστηκαν ε, ως ε, πιθανώς μολυσμένες. 2.300 περίπου τόνοι ζωοτροφής είχαν παραδοθεί σε περίπου 25 παρασκευαστές στη Γερμανία. Εκτός Γερμανίας δεν υπήρξε παράδοση 100 με 200 χιλιάδες τόνοι ζωοτροφών περιείχαν ο 2-10% ε, του πιθανός, ε, της πιθανώς μολυσμένης αυτής ουσίας είχαν ε, παραδοθεί σε περίπου 4.800 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Γερμανία. Ε, όμως ανιστάλλει πλήρως η εμπορική δραστηριότητα και η παράδοση και ό,τι πουλερικά, βοηδή. Σταμάτησε πλήρως η παράδοση. Αλλά σε κάποιες όρνηθες υπήρξε, για όρνηθες στη Γαλλία παραδείγματος χάρη υπήρξαν κάποιες ε, αποστολές. Μέχρι όμως ε, να ξεμπλοκαριστεί κάθε γεωργική εκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει καμία παράδοση από αυτήν. από τις 4.800 γεωργικές μεταλλές που έχουν μπλοκαριστεί, οι 939 για πουλερικά κυρίως, μεγάλες εγκαταστάσεις παραμένουν ακόμη μπλοκαρισμένες. Πάντως φαίνεται να μην υπήρξε εμπορία ούτε εξαγωγή μολυσμένων ζωοτροφών, με ελάχιστες εξαιρέσεις από τη Γερμανία. Τα τελικά αναλυτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε συμμόρφωση προ την κοινωτική νομοθεσία και γι' αυτό ε, βλέπουμε ότι το σύστημα ειχνηλασιμότητα είναι αποτελεσματικό. Θα εξακολουθήσουμε όμω να επαγρυπνούμε. Το ευτυχέ στην όλη κατάσταση είναι ότι τα παρατηρούμενα επίπεδα διοξίνη στι τροφέ όταν υπήρξε υπέρβαση του ορίου δεν ήταν πολύ ε, υψηλή υπέρβαση, άρα δεν υπάρχει κίνδυνο ε, για την δημόσια υγεία, για την υγεία των καταναλωτών από την κατανάλωση των ενδεχόμενη μολυσμένων ε, τροφών. Για μικρό βέβαια χρονικό διάστημα. Τι έχει κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο τη όλη κατάσταση. Οι υπηρεσίε μου είναι σε συνεχεί επαφέ με τι γερμανικέ αρχέ και άμεσα διέδισαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα κράτη-μέλη μέσω του ε, συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές. Ήταν επίσης επαφές με αρμόδιες αρχές σε τρίτε χώρες, δίνοντα τους μια σαφή εικόνα του συμβάντος σε όλους τους εμπορικούς μας εταίρους δώσαμε αυτή την ενημέρωση. Επίσης, οι αξιωματούχοι της Κομισιόν ήρθαν σε επαφή με τον κλάδο για να εξηγήσουν πώς μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο ο έλεγχος της παρουσίας διοξίνης στα τρόφιμα. Προσωπικά ήρθα σε επαφή με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Τροφίμων Γεωργίας Προσέσεις των Καταναλωτών της Γερμανίας, συγκεκριμένα την κυρία Άιγκνερ, στι 6 Δεκεμβρίου και ανταλλάξαμε απόψει για το τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθούν παρόμοια κρούσματα στο μέλλον. Σήμερα ήρθα σε επαφή με την Υπουργό, ε, τη Γερμανίδα, για μια ακόμη φορά, διότι με ανησύχησαν ε, οι ειδήσει του Σαββατοκύριακου ότι δεν δόθηκε πλήρης κατάλογος ε, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ενδεχομένω έχουν λάβει μολυσμένες ε, τροφές και δεν εδόθησαν ε, και οι σωστές πληροφορίες για την περιεκτικότητα της ουσίας σε συμπυκνωμένες τροφές. Πρόκειται για κάποιες εκατοντάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είναι μια σοβαρή παράβαση των διατάξεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει να πω ξεκάθαρο ότι οι γερμανικέ αρχέ έχουν δεσμευθεί πλήρω στην αντιμετώπιση ε, τη ε, μόλυνση αυτή. Θέλουν να το κάνουν αυτό αποφασιστικά και τάχιστα. Ενημερώθηκα ότι θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για τι δοκιμέ, θα δοθούν ακόμη περισσότεροι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο είναι σημαντικό οι ευρύτερε επιπτώσει για την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ζωοτροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπιστούν επίση κατεπηγόντω. Γι' αυτόν τον λόγο ε, μια ομάδα ε, του υπηρεσία τροφίμων ε, της ιατρικής υπηρεσίας θα επισκεφθεί τη Γερμανία σύντομα θα ενημερωθεί αλλά και θα ενημερώσει για, για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Οι γερμανικές αρχές είναι ενήμερες και έχουν συμφωνήσει να γίνει αυτή η επίσκεψη. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να στηριχθούμε στην πλήρη συνεργασία των γερμανικών αρχών. Θα συζητηθεί επίσης το ζήτημα αυτό και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας την επόμενη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου, στις Βρυξέλλες. Όπως προανέφερα, εξετάζουμε το ενδεχόμενο λήψη μέτρων και νομοθετικών μέτρων μεταξύ αυτών. Διότι το συμβάν αυτό κατέδειξε ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων ελέγχου που θα ε, εξασφαλίσουν, που θα εξασφαλίσουν και την αξιοπιστία των μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εξετάζουμε και το ενδεχόμενο σαφούς διαχωρισμού παραγωγή ζωοτροφών ή ουσιών που προορίζονται ε, για, ε, την, ε, για ζωοτροφές και όχι να τις αποσυνδέσουμε δηλαδή από τα λύπη και τις διάφορες άλλες που προορίζονται για τεχνικούς σκοπούς. Είμαι πεπισμένος και αισιόδοξο ότι με τα μέτρα όταν αυτά ληφθούν και εφαρμοστούν θα εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας. Thank you, Mr. Commissioner. Τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ντες θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση του σκανδάλου της διοξίνης στη Γερμανία. Εμένα με εξοργίζει ως αγρότη το ότι συνεχώς ε, πρέπει να ασχολούμαστε με τέτοια σκάνδαλα όπου από τη φαίνεται η ουσία είναι τσαπατσουλιά πιθανώς αλλά ίσως και εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε όσους νόμους θέλουμε στην Ευρώπη. Έχουμε στην Ευρώπη τους αυστηνότερους νόμους για τρόφιμα και ζωοτροφές. Έχουμε τις χαμηλότερες ουσίες ε, τα χαμηλότερα όρια με συγχωρείτε σε επικίνδυνε ουσίε και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλήρω αυτού του κινδύνου. Γι' αυτό θεωρώ πω θα πρέπει να είναι απέτηση και ε, γι' αυτό είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη. Πως όταν ο εισαγγελέα διαπιστώνει εγκληματική ενέργεια, οι ποινές να αυξηθούν κατά πολύ. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να τη γλιτώνουν με χρηματικές ποινές, πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή για να μην μπορούν να ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Χαίρομαι, κύριε Επίτροπε, για το ότι ήρθατε σε επαφή με τις γερμανικές αρχές και επισημάνατε πως θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Αυτή τη στιγμή παίζεται στη Γερμανία ένα πολιτικό θέατρο και δεν αντιμετωπίζεται σωστά η υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλοι μαζί το πώς θα συμπληρωθούν οι αυστηρές διατάξεις που έχουμε εκεί όπου αυτό χρειάζεται. Και πράγματι εδώ πέρα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Και μιλώ και εξ ονόματος της ομάδας μου, πως στην παραγωγή τροφίμων και λοιπόν προϊόντων θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός διαχωρισμός για να μην μπορούν να γίνουν τέτοιες επιμολύνσεις. Έχετε την υποστήριξή μας, λοιπόν κύριε Επίτροπε, για την βελτίωση των ε, ισχυουσών διατάξεων για να αποφευχθούν τέτοια σκάνδαλα στο μέλλον. Τώρα για την ομάδα <clears throat> Σοσιαλιστών Δημοκρατών, η κυρία Ρόντους, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκπλήσω με αυτά τα οποία είπατε. Αλλιώς θα λέει ο τύπος, στη Γερμανία τουλάχιστον. Και εμένα με εξοργίζει το ότι προκύπτουν συνεχώς σκάνδαλα στον τομέα των τροφίμων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Γνωρίζω πως ο κανονισμός και οι νόμοι δεν μπορούν να εμποδίσουν από μόνα τους εγκληματικές δράσεις. Αλλά πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τιμωρηθούν όσο το δυνατόν σκληρότερα και να γίνει όσο το δυνατόν δυσκολότερο το έργο των υπευθύνων. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αντιμετωπίζεται με τα συνήθη μέσα τέτοια εγκληματική δράση στον τομέα των τροφίμων. Επίσης, συχνά βλέπετε πως οι χρηματικές ποινές είναι τόσο χαμηλές που χρηματοδοτούνται από τα τρέχοντα της ε, επιχείρησης, τα τρέχοντα έξοδα. Επίσης, αποδείχθηκε εδώ πέρα πως η αρχή του αυτοελέγχου έχει πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει η αρχή του ο υπεύθυνο πληρώνει ή εν πάση περιπτώσει είναι και ποινικά υπεύθυνο σε ολόκληρη την αλυσίδα των τροφίμων. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται επίσης οι αθώοι και να πληρώνουν οι άνθρωποι που είναι παρακάτω στην αλυσίδα και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να αποζημιωθούν και από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει. Εδώ πέρα πρέπει να το δούμε ευρωπαϊκά το ζήτημα τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται συνεχώς στον τομέα της ασφάλειας των ε, τροφίμων ξεκαθαρίζουν ένα πράγμα. Πρέπει να δούμε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών και να υπάρχει πλήρης ίχνη λασιμότητα. Εδώ πέρα πρέπει να βελτιωθεί και η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο θα πάρει για την ομάδα των φιλελευθέρων η κυρία Λεπάζ για δύο λεπτά παρακαλώ. Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτή σας τη δήλωση. Γνωρίσαμε τέτοιου είδους επεισόδια σε μια δεκαετία στην Ευρώπη και πρέπει να χαιρόμαστε ότι το σύστημα συναγερμού λειτουργήσε όμως είναι απαράδεκτο ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Η υγεία των καταναλωτών των Ευρωπαίων δεν μπορεί να είναι η μεταβλητή προσαρμογή ενός συστήματος που ε, προωθεί την μείωση του κόστους και είναι μια έμεση ενθαρρύνση ε, όταν επιβάλλονται πολύ χαμηλές ποινές. Και ξέρετε κύριε Επίτροπε, για να έχουμε εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Τι δράση έχετε υπόψη σας να αναλάβετε. Χαίρομαι που προηγουμένως αναφερθήκατε στο ότι θα υποχρεώσετε να γίνει διαχωρισμός της χρήσεως προετοιμασίας των βιομηχανικών λοιπόν και των λιπαρών ουσιών που πηγαίνουν για την κατανάλωση. Είναι μια υποχρέωση και δεν είναι μια δυνητική ευχέρεια στην όλη διαδικασία της παρασκευής των προϊόντων αυτών, τόσο ώστε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα. Ε, δεύτερον, είναι ασύνηθες η να διοργανώνεται έτσι η φερεγγιώτης. Τι δράσεις θα εφαρμόσετε κύριε Επίτροπε, ούτω ώστε να μπορείτε να εγγυηθείτε ότι τέτοιες ε, πράξεις θα παραμένουν, δεν θα παραμένουν ατιμόρυτες, διότι η υπευθυνότηση είναι η μεγαλύτερη ασφάλιση. Μετά, τι δράση θα ακολουθήσετε για να βελτιώσετε την εποπτεία που εφαρμόζουν τα κράτη. Πέρασαν περίπου τις εβδομάδες από τη στιγμή που δόθηκαν αυτά τα λιπαρά και που χτύπησε ο συναγερμό. Ε, δεν φταίει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό, αλλά είναι ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές αυτό. Νομίζετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά αυτό το στοιχείο, κύριε Επίτροπε. Σα ευχαριστώ. Σας πολύ, κύριε Λεπάζ. Ο κύριο Χάουσλινγκ για δύο λεπτά έχει το λόγο την ομάδα Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, διαπιστώνουμε πως η εμπιστοσύνη του καταναλωτή κλονίζεται πάλι και αναρωτιέται ο καταναλωτής τι κάνουν οι εθνικές αρχές, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση. Οπότε, κύριε Επίτροπε, θεωρώ πως αυτό δεν ήταν ένα περιστατικό ή μία σύμπτωση, νομίζω πως συγκεκριμένες επιχειρήσεις κερδίζουν εκατομμύρια με την ε, ανάπτυξη αυτών των ε, ουσιών και τελικά την πληρώνει η αγρότη του δεν τίποτα και ο καταναλωτή. Οπότε νομίζω πω εδώ πέρα ο έλεγχο είναι σε λάθο σημείο. Υπάρχουν μία χούφτα επιχειρήσει που εργάζονται στη Γερμανία με τα λύπη. Γιατί δεν κάνετε πιο στοχευμένου ελέγχου σε αυτέ. Και περιμένουμε συμπτωματικά ε, να ανακαλύψουμε κάτι και να τρέχουμε εκ των υστέρων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ανάλυση που θα βασίζεται σε μια επιτήρηση που θα βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου. Και το θέμα εδώ πέρα είναι τι κάνει η ΕΦΣΑ. Είναι γερμανική η περίπτωση ή υπάρχουν και άλλε περιπτώσει στην Ευρώπη που πιθανώ δεν έχουν ανακαλυφθεί. Θεωρώ πω εδώ πέρα συμφωνούμε, χρειαζόμαστε έναν θετικό οριστικό κατάλογο για το τι επιτρέπεται να μπει στι ζωοτροφέ. αυστηρή διαδικασία διοδότηση των επιχειρήσεων και βεβαίω οπωσδήποτε χωριστά ρεύματα παραγωγής. Αλλά χρειάζεται ανακατεύθυνση βασική της πολιτικής. Γιατί τελικά τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τρώνε το φαΐ τους τα ζώα στο χωράφι και όχι να είναι βιομηχανικό προϊόν και να ψάχνει να το αγοράσει από κάποια επιχείρηση ο αγρότης. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η ε, γεωργική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει γιατί τελικά ολόκληρη η γεωργία υφίσταται τη ζημιά κάποιων εγκληματιών εδώ πέρα. Ε, αυτό πρέπει να εμποδίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα την θέση πολλών Γερμανών γεωργών. Ε, δείχνω κατανόηση για τη θέση στην οποία βρίσκηκαν οι Γερμανοί γεωργοί τέτοια εποχή. Εδώ και τρία χρόνια στη Βόρεια Ιρλανδία είχα αυτή την εμπειρία όταν περάσαμε πολύ παρόμοια περίοδο και πρόβλημα. Και πρέπει να πω ότι αυτοί υποφέρουν πραγματικά, οι γεωργοί υποφέρουν πραγματικά. Αυτοί που επουδενή, υπό οποιαδήποτε μορφή δεν αναμειγμένοι σε αυτά τα γεγονότα. Αναφέρθηκε η λέξη εγκληματική στην ενέργεια. Εκείνοι που είχαν εγκληματική πρόθεση είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα και έχουν ανακατευθεί. Και θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί το κάνουν. Και πρέπει να σα πω, Επίτροπε, το κάνουν για να βγάλουν πολλά λεφτά, να βγάλουν μεγάλα κέρδη. Αν πρόκειται περί αυτού, θα πρέπει να διωχθούν. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι εκεί αυτοί που παράγουν τα τρόφιμα που είναι υπεύθυνοι. Είναι εκείνοι που δίνουν τι ύλε εκείνου που παράγουν τι ζωοτροφέ που είναι υπεύθυνοι. Και θα πρέπει να κινηθούμε κατά αυτόν, ούτω ώστε να μην ξανασυμβεί και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Διότι μπορώ να καταλάβω πολύ καλά γιατί οι καταναλωτέ ε, κλονίζονται, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του. Διότι όπω είπε και κάποιο, αυτό συνέβη ξανά και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αλλά μην το εξετάσουμε σφαιρικά με ολοκένουργια νομοθεσία. Σε εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουίλς για δύο μισή λεπτά από την ομάδα της αριστεράς. Das sind die drei... Κοιτάξτε, ε, άλευρα, και οι λιπεσουσίες είναι η αλυσίδα των ζωοτροφών στην ε, Γερμανία και είχαμε πάρα πολλά τέτοια σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια. Το θέμα εδώ πέρα δεν είναι η εθνική ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν το ζήτημα είναι να έχουμε μεγάλα κέρδη με φθηνές ζωοτροφές. Ο ανταγωνισμό στον τομέα των ζωοτροφών ε, είναι πάρα πολύ σκληρό στη Γερμανία για να επιτευχθούν οι χαμηλότερε ε, τιμέ και βεβαίω θα πρέπει να είναι πρέπει να είναι όσο δυνατόν φτηνότερες οι ζωοτροφέ. Η δε έλεγχη είναι ελάχιστη. το κράτος βασίζεται όλο και περισσότερο στον αυτοέλεγχο των ε, παραγωγών και έχει κάνει οικονομίες στο εξειδικευμένο προσωπικό. Υπ' αυτές τις συνθήκες λοιπόν μπόρεσαν να φτάσουν από την παραγωγή βιοντίζελ ε, οι μολυσμένες ε, διοξίνες στην αλυσίδα των ζωοτροφών. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει εμποδιστεί κάτι τέτοιο εάν ρεύνοταν ε, ε, αυτή η ουσία πριν καταλήξει στα συστατικά της ζωοτροφής. Τώρα λοιπόν θα έχουμε πάλι αμέτρητους καταναλωτές οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με διοξύνη 80% της διοξίνης την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος προέρχεται από τις ζωικές τροφές, δηλαδή αυγά, γάλα, κρέας. Η Food Watch, η οργάνωση, απαιτεί να υποχρεωθούν οι παραγωγοί να ε, αναλύουν κάθε φορτίο για διοξίνη και PCB πριν το βάλουν, το αναμίξουν με τα υπόλοιπα συστατικά. Δεν θα επιτρέπεται να μπαίνει κανένα τέτοιο φορτίο πριν αναλυθεί και βεβαίως τα επιβαρημένα θα πρέπει να καταστρέφονται. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε ε, τυχόν ε, χρήση αυτών των ουσιών. Επίσης θα πρέπει και τα εργαστήρια να είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν υπερβάσεις των ορίων αυτών στις αρμόδιες αρχές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει για το κρέας ίχνη λασιμότητα. Τα δε τωρινά και προηγούμενα σκάνδαλα στη Γερμανία έδειξαν πως ο έλεγχος ρουτίνας του κράτους είναι οπωσδήποτε απαραίτητος. Πώ θα το εφαρμόσετε λοιπόν αυτό και πώ θα το επιβάλλετε κύριε Επιτροπή. Ο κύριο Πάσκα, ο επόμενο εγγεγραμμένο ομιλητή εκ μέρου τη Ευρώπη Ελευθερία Δημοκρατία, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα. Οπότε θα συνεχίσουμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Ο κύριο Λίζε θα πάρει λοιπόν το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταναλωτέ και γεωργοί θα πρέπει να προστατευθούν από τους ανεύθυνους αυτούς εμπόρους. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησαν οι συνάδελφοι για τη Γερμανία, αλλά δυστυχώ είχαμε τέτοια σκανδαλά και σε άλλε χώρε στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα, ο εισαγγελέα θα ερευνήσει τι ποινικέ ευθύνε και ελπίζω οι Γερμανοί εισαγγελεί και όσοι αναμειχθούν και από άλλε χώρε αναφέρθηκε και η Ολλανδία ως κομμάτι της αλυσίδας, να εργαστούν γρηγορότερα από τους Ιρλανδούς εισαγγελείς, όπου τώρα καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο του 2008. Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα αυτή τη φορά. Και να σας ζητήσω το σκάνδαλο αυτό να το δούμε σωστή του διάστοση. Μιλάμε για τέσσερις φορές πάνω από το όριο, κάτι το οποίο είναι κακό γιατί οπωσδήποτε το όριο υπάρχει εκεί για κάποιο λόγο. Αλλά οπωσδήποτε το όριο το έχουμε επιλέξει κατά τρόπον ώστε να φτάσουμε σε μακροπρόθεσμη ζημία όταν το ξεπεράσουμε κατά 100 φορές. Οπότε δεν μιλάμε για οξύ κίνδυνο, μιλάμε για πρόληψη. Και μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο την τελευταία φορά είχαμε φτάσει 700 φορές πάνω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πράγματι βλέπουμε εδώ πέρα πως υπάρχει και μην ξεχνάτε μείωση κατά το 1 δέκατο με την ε, νομοθεσία περί αποτέφρωσης. Όμως χρειάζονται πράγματι μέτρα πανευρωπαϊκά, χρειάζεται παρακολούθηση των ε, διοξινών, διαχωρισμός των λοιπόν, χρειάζεται θα έλεγα ένας νόμος καθαρότητας ανάλογος με αυτό της μπύρας για τις ζωοτροφές και να δούμε βεβαίω οπωσδήποτε και του ανθρώπου οι οποίοι έκαναν αυτέ τι ε, εγκληματικέ συνελήψει για να μην συμβαίνουν συνέχεια τα ίδια πράγματα. Ε, για ένα λεπτό ο κύριο Κάπουλα Σάντο θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορούμε παρά να το επαναλαμβάνουμε το ότι η Ευρώπη έχει την πιο αυστηρή νομοθεσία από ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και δεν μπορούμε αυτή την εικόνα να την αμαυρώσουμε επουδενή. Αυτό θέλουν οι καταναλωτές μας και οι αγορές τις οποίες εξάγουμε επίσης. Και τεράστια δουλειά έχει γίνει από τους παραγωγούς όσον αφορά τις επενδύσεις για να βοηθήσουν να πετύχουν αυτό το στόχο. Εάν ε, το πρόσφατο αυτό γεγονός που συνέβη στη Γερμανία είχε συμβεί κάπου αλλού στον κόσμο, ίσως να μην το είχαμε ακούσει καν. Συνέβη όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που συνέβη στη Γερμανία είναι απαράδεκτο βέβαια και θα πρέπει να εξεταστεί και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ακριβώς τι συνέβη και να βρούμε ποιος είναι υπεύθυνο. διότι πρόκειται περί εγκλήματος. Δεν είναι απλώς ένα συμβάν δεν έχει ανακαλυφθεί από πού προήρθε η επιμόλυνση και θα αυτό με εκπλήσει ούτε ε, έχει διελευκανθεί ποια είναι η ευθύνη των γερμανικών αρχών, δηλαδή που υπήρξαν ελλείψεις όσον αφορά τους ε, ελέγχους. Αυτό το θέμα δεν έχει εξεταστεί και η σοβαρότητα της καταστάσεως σημαίνει ότι θα πρέπει να, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει αντικειμενικά. Ευχαριστώ. Κυρία Ρέιμερς, για δύο λεπτά παρακαλώ θα πάρει το λόγο τώρα. Ε, Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με το περιστατικό αυτό δεν μιλάμε μόνο για ένα σκάνδαλο. Βλέπουμε την εικόνα μας στον καθρέφτη. Πόσο καιρό λέμε πως η Γεωργία πληρώνει ένα πάρα πολύ υψηλό τίμημα μέσω του έντονου αυτού ανταγωνισμού. Ο αγώνας πλέον δεν είναι μόνο για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, είναι κάτι το παραπάνω. Και άρα πολύ όλο και περισσότεροι ακολουθούν όλο και συχνότερα εγκληματικέ μεθόδους. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να περάσουμε περισσότερους νόμους, περισσότερους ελέγχους με μεγαλύτερο κόστος. Μπορούμε να επιβάλλουμε αυστηρότερες ποινές. Τίποτα από αυτά δεν θα σταματήσει την εγκληματική ενέργεια ενός τέτοιου ολοκληρωτικού αγώνα. Πρέπει να δούμε την ουσία του κακού, την αιτία. Δηλαδή ότι θέλουμε όλο και περισσότερα, όλο και φθηνότερα. Ως γεωργός και εγώ έχω ζήσει την αδυναμία ε, να αντιμετωπίσω τέτοιους ε, ανθρώπους. Και έχω ζήσει το πώς είναι να είναι κανείς αθώος και να εμπλέκεται σε μια τέτοια υπόθεση. Γι' αυτό ρωτάω την Κομισιόν τι θα κάνετε εσείς και οι συναδελφοί σας για να έχουν πάλι προσθέμενη αξία τα τρόφιμα. Χαιρετίζω τις προτάσεις σας αλλά δεν θα λύσουν το βασικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Στάς για ένα λεπτό, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, το σκάνδαλο αυτό έχουν εντύπωση δηλαδή πως το έχουμε ξαναζήσει. Γιατί η κρίση είναι ίδια όπως και πριν από 12 χρόνια στο Βέλγιο. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δείχνουν πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον τομέα των ε, ζωοτροφών που δεν έχουν καθόλου συνείδηση και είναι διατεθειμένοι να κάνουν εγκληματική απάτη εις βάρος των αγροτών και της υγείας των καταναλωτών και αυτό είναι αδιανόητα. Οπότε χρειάζεται σήμερα να γίνει ένα είδος stress test της νομοθεσίας κάτι το οποίο ζητάμε από το Συμβούλιο Γεωργίας αλλά χρειάζεται και έλεγχος. Υπάρχει αυτό έλεγχος στον κλάδο αλλά πέρα από τον αυτοέλεγχο πρέπει να υπάρχουν περισσότερες αυστηρότε περισσότεροι αυστηρότεροι έλεγχοι από τις εθνικές αρχές με σωστή αναλογία και δεύτερον θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει περισσότερος έλεγχος από την υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικής στην Ιρλανδία έλεγχος του ελέγχου. Διάβασα πως τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει τρεις αποστολές από τον FBO. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να δώσετε οδηγία στον, ε, στο Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικής να κάνει περισσότερα πράγματα για το ζήτημα των διοξινών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα, ο οποίος ο, ο, ήταν ομιλητής εκ μέρους της Ευρώπης της Ελευθερίας Δημοκρατίας, είναι στην αίθουσα και θα του δώσω το λόγο για δύο λεπτά όπως έχει προδιαγραφεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς κανόνες, κανονισμούς ε, που βεβαίως ε, στόχο έχουν να βελτιώσουν ε, την ποιότητα των τροφίμων. Πάρα πολύ υπάλληλοι, θεσμικά όργανα, οργανισμοί υποτίθεται πως αγγιούνταν μία ποιότητα των τροφίμων. Όμως βλέπουμε τώρα πως ε, έχουν πάλι τα πράγματα. Η Ευρώπη πάλι αντιμετωπίζει δηλητηριώδη τρόφιμα και δεν ξέρει ε, ο γραφειοκρατικός μηχανισμός τι να κάνει. Για να περιγράψω καλύτερα την ε, κατάσταση, ας δούμε τι κοκτέιλ έχουμε μπροστά μας. Οι διοξίνες είναι από τις πιο επικίνδυνες ουσίες που έχουν παραχθεί ποτέ από τον ε, άνθρωπο. Είναι επικίνδυνες για τα κύτταρα, για την ανάπτυξη. Αυξάνουν το ποσοστό θνησιμότητας ε, και διαταράσσουν τη ροή των όρμονων. Έχουν σορευτική επίδραση ε, στον οργανισμό και Ξέρετε πως ποσότητα διοξίνης ίση με τον κόκο ενός ρυζιού μπορεί να δηλητηριάσει ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Η εταιρεία Hannes Jens ε, της ε, Γερμανίας από το Μάρτιο 2010 είχε διακινήσει 3.000 τόνους λίπη μολυσμένα με διοξίνη και είχαν πάει προς Ολλανδία και Δανία. Έρωτο, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση που παραδίδει ύλες σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις να μην είναι καταγεγραμμένη. Τι κάνουν οι αρχές στη Γερμανία εάν είναι δυνατόν χωρίς έλεγχο να λειτουργεί κανείς. Τι, τι, τι γίνεται με το κτηνιατρικό έλεγχο από το Μάρτιο του 2010 μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να διαπιστώσει την ε, μόνηση αυτή. Και τι θα γίνει και με την τελική καταστροφή αυτών των ε, τροφίμων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενος ο κύριος Βόιτσεχόφσκι για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο αλλά λίγα λέω. Είναι μεγάλη απειλή για χιλιάδες ανθρώπους, απειλή για την υγεία, απειλή για τη ζωή τους. Και ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Πάντως αυτή η περίπτωση θα πρέπει να δούμε τι γεωργία έχουν, να μας κάνει να σκεφτούμε τι γεωργία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωργία έχει γίνει βιομηχανία. Το κρέας ε, παράγεται σε τεράστιες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε επίσης τη βιομηχανία των ζωοτροφών, όπου τα ζώα ταΐζονται με τροφές που είναι μολυσμένες με διοξίνη ή με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και δεν λειτουργεί αυτή η κατάσταση, δεν εγγυάται την ασφάλεια των τροφίμων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στα αγροτικά που είχαμε πριν από χρόνια, στην Πολωνία, όπου η παραγωγή των ζωοτροφών γινόταν εκεί, επί τόπου. Ευχαριστώ κυρία Λιωτάρ για ένα λεπτό. Eh, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το Μάρτιο του 2010 γνώριζε η, η υπεύθυνη επιχείρηση πώς ήταν μολυσμένο το προϊόν. Πώς είναι δυνατόν να μην ε, προέκυψε αυτό σε κανέναν δημόσιο έλεγχο από τις ε, κρατικές αρχές. Επαρκούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Προφανώς όχι, αλλιώς θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει αυτή την ε, κρίση. Διατροφικά σκάνδαλα συμβαίνουν. Σκεφτείτε πέρα από τη διοξίνη και τα προϊόντα από κλόνους που είχαν καταλήξει στα καταστήματά μας πέρσι. Πρέπει λοιπόν να γίνονται οι έλεγχοι καλύτερα και συχνότερα και οπωσδήποτε θα πρέπει το αποτέλεσμα αυτών ελέγχων να είναι δημόσιο. Μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων και της υγείας των πολιτών μας. Επιπλέον, απευθύνω έκκληση στην ε, Κομισιόν να στηρίξει τους αγρότες εκείνους οι οποίοι έπαθαν όσον αφορά την αποζημίωσή τους. Ευχαριστώ και τον λόγο τρέχει ο κύριος Σάκνιο για ένα λεπτό. Thank you, President. <clears throat> First, may declare an interest. I am... Κοιτάξτε, είμαι παραγωγός ο ΟΟΝ, Βρετανός. Η, η μόλυνση της διοξινή φαίνεται ότι οφείλεται στην αποτυχία στο να μην ακολουθηθούν οι πιο ψηλέ ε, προδιαγραφές για την επεξεργασία ζωοτροφών. Ακολουθήθηκαν διαδικασίες ε, για την παραγωγή βιοκαυσίμων ανταυτού από, από κράμβη, από σπόρους κράμβης. Λοιπόν, όλο αυτό είχε δεινέ συνέπειε, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέμα μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν χρειάζεται παραπάνω νομοθεσία. Οι Γερμανοί εντοπίσαν το πρόβλημα. Μα το έκαναν τα δέοντα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε σύστημα ασφάλισης, αν θέλετε, που καλύπτει και την παραγωγή ζωοτροφών και την παραγωγή των αυγών. Άρα είναι απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη στη Γερμανία. Λοιπόν, αν επιμένετε για πολύ καλά αυγά, ζητήστε το Lion. Λοιπόν, σας δώσουμε με σύμβολο το λεοντάρι και οι Βρετανοί παραγωγοί τα χάρη σας δώσουν τέτοια αυγουλάκια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Αν μιλάμε σήμερα για κρίση, αυτό γίνεται γιατί τέλος πάντων το σύστημα παρόλα αυτά λειτουργήσε. Έχουμε ένα σύστημα προστασίας των καταναλωτών με τα υψηλότερα ανά τον κόσμο πρότυπα Άρα πρέπει ε, να ε, το έχει υπόψη το αυτή τη στιγμή αυτό ο καταναλωτή. Βέβαια, το σύστημα δεν λειτουργήσε σωστά. Πριν όμως προχωρήσουμε σε ένα νέο σύστημα, θα ήταν καλύτερα, κατά την άποψή μου, να διερευνήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση ανακάλυψης του προβλήματος και θα πρέπει να διερωτηθούμε για τα αίτια αυτής τη καθυστέρηση. Πρέπει όμως ακόμη, κατά την άποψή μου, να διερωτηθούμε για το γιατί. Ναι, με να καταγγείλουμε την εγκληματική πράξη, αλλά νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει ο γεωργικός ε, κόσμος ε, έναν αγώνα για όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές ε, στις πρώτες ύλες. Δύο σε συμπεριφορές που δεν είναι χαρακτηρίσιμες, δεν είναι σωστές. Θα εξετάσετε λοιπόν το ενδεχόμενο αύξηση των ποινών και προστήμων για τέτοιου είδους ενέργειες. Και δεύτερο ερώτημα, πώς εμείς μπορούμε να στηρίξουμε άμεσα, άμεσα το επαναλαμβάνω, τους κτηνοτρόφους που πλήττονται, διότι είναι τόσο μικρά τα περιθώρια που αν κάποιοι δεν έχουν στήριξη άμεσα, έστω και μια προκαταβολή των ποσών που τους οφείλονται, όταν θα έχει καταλήξει η διαδικασία θα έχουν εξαφανιστεί αυτή η παραγωγή αν ακολουθήσουμε την κανονική ταχύτητα. Ευχαριστώ. υπάρχει ένα ερώτημα προς τον ομιλητή. Έχετε ερώτηση. Κύριε Ομπερμάιρ, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να απευθυνθώ λοιπόν στον προλαλήσαντα είπε πως κατά βάση λειτουργεί το σύστημα. Ξέρετε, δεν το ανακάλυψε το σύστημα. Οι καταναλωτές βοήθησαν στην ανακάλυψη. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν ξέρετε πως υπάρχουν μελέτες που λένε πως είναι διατεθωμένοι να πληρώσουν παραπάνω οι καταναλωτές εάν ξέρουν πως θα είναι τα προϊόντα πιο ποιοτικά και ε, με καλύτερε συνθήκε για τα ζώα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Ακούστε, νομίζω ότι ο συνάδελφο που έθεσε το ερώτημα, ουσιαστικά σχόλιο ήθελε να κάνει, σχόλιο για την κατάσταση και όχι να μου θέσει ένα ερώτημα. Φυσικά και γνωρίζουμε, πώς να το πω, ότι ε, το σύστημα ε, δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά Έχουμε ένα πολύ σοβαρό σύστημα. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι δεν γίνεται τίποτα, ενώ έχουμε τα αυστηρότερα, τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε στον κατάλογο. Ο κύριος Ντεκάστρο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ και εγώ πάνω απ' όλα τον Επίτροπο mm. που ήρθε εδώ σήμερα στην Ολομέλεια και αναφερθεί σε αυτή την υπόθεση που ανησυχεί του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Την επόμενη εβδομάδα και η Επιτροπή Γεωργία, τη οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, θα εμβαθύνει στη συζήτηση όσον αφορά τι συνέπειε αυτού του σοβαρού επεισοδίου. Παρότι ότι η Ευρώπη κάνει πολλέ προσπάθειε όσον αφορά την ευστιστική ασφάλεια, χρειάζονται και άλλε προσπάθειε όσον αφορά τη διαφάνεια και του ελέγχου για να αποφευθούν και άλλε παρόμοιε υποθέσει ε, μολύνσεω στα τρόφιμα. Υπενθυμίζω τελευταίο χρόνο το Κοινοβούλιο θέτησε μια έκθεση πρωτοβουλία σχετικά αφορά την ποιότητα των γεωρικών προϊόντων και κυρίω αυτή η Ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση οθέτησε τον κανονισμό για τι πληροφορίε που δίδονται στου καταναλωτέ στο φάρτο τρόφιμα και υποχρεωτικέ ενδείξει στην ετικέτα του τόπου προέλευση των γεωρικών προϊόντων. Σημαντική καινοτομία που δυστυχώ όμω σταμάτησε στου 8 ε, Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Υγεία. Εμεί στη δεύτερη ανάγνωση προσπαθούμε να την επανεισαγάγουμε διότι είναι σημαντική, ε, σημαντικό μέτρο για τη διαφάνεια και προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται προ σωστή κατεύθυνση δείχνοντα ότι είναι με το μέρο των καταναλωτών. Ελπίζουμε και την πλευρά του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τοποθέτηση θα είναι ανάλογη. Ευχαριστώ. ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, όπως ήδη ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι, ε, και εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτά που ποιόθηκαν, ότι η παρούσα νομοθεσία, η νομοθεσία της Ευρώπης, σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί. Δεν έγκυται εδώ το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα έγκυται στην εφαρμογή των νόμων στους ελέγχους και το σύστημα των κυρώσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν θεσπίζουμε εμείς νόμους χωρίς σύστημα κυρώσεων το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να εφαρμόσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως τότε θεσπίζουμε νόμους οι οποίοι νόμοι δεν θα έχουν αποτελέσματα. Αναφέρθηκε κάτι σημαντικό. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για τον κανονισμό που στηρίζει τον, την όλη προσέγγιση για τις ζωοτροφές και έπρεπε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ πρώτων υλών, να γίνεται διαχωρισμός πρώτων υλών για τις ζωοτροφές και ε, των λοιπόν λιπαρών ουσιών που πηγαίνουν για τεχνικές κατεργασίες. Είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε τον διαχωρισμό και εγώ πριν από 10 χρόνια είχα προτείνει όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν ύποπτη προέλευση θα έπρεπε ε, να, να μην χρησιμοποιούνται, να απαγορεύονται. Διότι εγώ λυπάμαι τους γεωργούς που επανειλημμένα πλήττονται από αυτή την μόλυνση και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ροντσούλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να είμαι μία από εκείνου που θα υπέγραφε εκείνη την ερώτηση, διότι θεώρησα ότι είναι θεμελιώδε αυτό μετά από αυτά που συνέβησαν τι τελευταίε εβδομάδε. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε η συζήτηση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Πότε είναι υγιή τα τρόφιμα παράγονται που καθημερινά καταναλώνονται από εκατομμύρια ε, Ευρωπαίους καταναλωτές. Είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα που έχουμε στο τραπέζι μα είναι ασφαλή. Η ποιότητα των πρώτων υλών είναι θεμελιώδου σημασία για να μπορούμε να εγγυθούμε την αυθεντικότητα του τελικού προϊόντο. Έλεγχο συνεχή από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι είναι ο μόνο τρόπο για να αποφύγουμε την επιμόλυνση των τροφίμων και να μπορούμε αμέσω να εντοπίσουμε ενδεχόμενου κινδύνου. Το νέο επεισόδιο στη Γερμανία δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα και για τα μεταποιημένα προϊόντα η ένδειξη προέλευση στην ετικέτα όπω ήδη υπογραμμίστηκε και από την συνάδελφο Ντεκάστρο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτού, να μπορεί να ξέρει ο καταναλωτή την προέλευση κάθε προϊόντο το οποίο αγοράζει και η ασφάλεια των τροφίμων των προϊόντων αυτών μπορεί να την εγγυηθούμε μόνο αν υπάρχει κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή. Ήδη προβλέπει νομοθεσία διαδικασίε και ελέγχου, ούτω ώστε να έχουμε την εγγύηση ότι το τρόφιμο που φτάνει στο τραπέζι μα είναι ιδεώδε για κατανάλωση και ότι οι κίνδυνοι για τη μόλυνση στο ελάχιστο. Αλλά ο στόχο μα θα πρέπει να είναι τώρα να συμβάλλουμε καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ε, των προϊόντων. Υπογραμμίζω με περηφάνεια ότι αύριο το Ιταλικό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ένα νόμο που επεκτείνει την ένδειξη προέλευσης και την καθιστά υποχρεωτική για όλα τα τρόφιμα ε, που σήμερα δεν έχουν αυτό το σήμα και την αναφορά. Η προέλευση των προϊόντων όπως είναι το χείριο κρέας και όπως είναι και το γάλα μακράς διαρκείας, τα οποροκυπευτικά και κάποια προϊόντα όπως η πορτοκαλάδα τα χρειάζονται αυτά. Ελπίζω να εμπνευστεί από αυτή την νομοθεσία η Ευρώπη και εγώ θα παρεύω για να προσπαθήσω να πετύχω μεγαλύτερη ε, ενημέρωση, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτού, μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι μέσα αυτά τα οποία θα ευνοήσουν μια υγιή και πραγματική αυθεντική ε, διατροφή. Ευχαριστώ. Κύριος Ουλσκοφ. Η κυρία Ουλσκοφ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Το σημαντικό θέμα είναι πώς να αποφύγουμε νέα σκάνδαλα και νέους ε, κινδύνους. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισκεφθεί ε, τη Γερμανία και ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα συζητήσει το θέμα. Θα ήταν σκάνδαλο αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο, ήταν σκανδαλώδες. Διότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ, θα πρέπει να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις, πράγματι. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και καλύτερα, κυρώσει. μεγαλύτερες κυρώσεις. Και θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να διενεργούν τους ελέγχους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Όμως τελικά έτσι θα αποφύγουμε τη μόλυνση των τροφίμων και να αποφύγουμε και τη μόλυνση των τροφίμων που καταναλώνει ο άνθρωπος. Ως καταναλωτές δεν θέλουμε να τρώμε μολυσμένο φαγητό και θα πρέπει οι καταναλωτές να ξέρουν ότι είναι σίγουροι αυτό που τρώνε ότι είναι υγιές. Ευχαριστώ. Η κυρία Παρβανόβα έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συναδελφέ. Αυτό που συμβεί τον Δεκέμβρη στη Γερμανία και αυτό που οι υπηρεσίε, όχι μόνο χιλιάδε κανοντές έθεσε σε κίνδυνο αλλά επίση έδειξε το πόσα παραθυράκια υπάρχουν στο σύστημα. Είναι παραπάνω σχετικό το ότι οι γερμανικέ αρχέ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσαν να πάρουν ότι τίποτε από τα μολυσμένα δεν θα μπορέσει να μπει στην αλυσίδα τη διατροφική, δεν θα μπορέσει να αποτελεί, να αποτελεί συστατικό αυτόν που τρώμε. Επομένω, αυτό είναι ένα βάρο από την άλλη μεριά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για κατάσταση ανάγκη που συζητούμε σήμερα. Και άρα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα πρέπει αυτό να αποτελεί προεπιτούμενο για να προστατεύει η υγεία του καταναλωτή. Διότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα επιβεβαιώσουν ότι τίποτε από τα μολυσμένα δεν πήγε στην τροφική αλυσία Ούτε ω μεταποιημένο. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία ε, ε, έλαβαν ή έπρεπε να λάβουν υπόψη ισχύει ότι θα υπάρξει ενημέρωση καταναλωτών στο μέλλον για να αποσοβηθεί άλλη τέτοια τροφική κρίση. Ευχαριστώ. Κυρία Κέστιγκερ για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν οδηγηθεί σε αβεβαιότητα μέσω του σκανδάλου αυτού όσον αφορά ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων σε τελική ανάλυση έχει βλεφθεί η διεθνής εικόνα της Γεωργίας μέσω κάποιων ανθρώπων που επέδειξαν κάποια μελή συμπεριφορά. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων. Επίσης θα πρέπει και αυτό είναι μόνο η αρχή να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Θα πρέπει να ληφθούν επίσης άμεσα μέτρα για να σταματήσουν και να μην είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες πρακτικές. Επίσης, αντιλαμβάνεστε πως δεν έχουν καμία θέση βιομηχανικά απόβλητα στην ε, αλυσίδα των ε, ζωοτροφών. Δεν είναι δυνατόν καν να έχουμε τέτοια επιμόλυνση των ζωοτροφών. Είναι λοιπόν απαραίτητος, απαραίτητος ο έλεγχος τέτοιων επιχειρήσεων γιατί δεν είναι δυνατόν να αποδεχτεί ο αγρότης ο οποίος ελέγχεται πολλές φορές μες στο έτος οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν τις πρώτες ύλες να μένουν ανεξέλεγκτες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε όμως πώς αντέδρασαν τελικά σωστά οι αρμόδιες ε, αρχές. Επίσης χρειάζονται στήριξη οι αγρότες οι οποίοι έχουν πληγεί χωρίς να φταίνε χιλιάδες αυτή τη στιγμή αγρότες απειλούνται με χρεοκοπία και αντιλαμβάνεστε πως αυτή τη στιγμή ε, στον τομέα των χοιρινών προϊόντων τιμή του παραγωγού είναι γύρω στα 20 cents το κιλό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πως εδώ πέρα η κατάσταση επιδεινώνεται από το ότι αυξήθηκε και το κόστος της ε, παραγωγής και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν επιτρέπεται να κλονίζεται για λόγους κερδοσκοπίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα η κυρία Στάιλερ για ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, η διοξίνη είναι ένα πολύ επικίνδυνο χημικό γνωστό ως καρκινογενές. Ε, όταν κατά λάθο χρησιμοποιηθούν τέτοια ε, υλικά για την κατασκευή μέσα στην αλυσίδα κατασκευή ζωοτροφών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. 77 φορές παραπάνω από το εγκεκριμένο ποσοστό διοξίνη περιείχαν αυτά τα τρόφιμα. Ακριβώς γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι για να αποφύγουμε να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές από τέτοιου είδου ε, μολύνσει. Ε, μόνο που μέχρι να γίνει ο έλεγχο, είχαν φτάσει τα προϊόντα αυτά σε όλα τα μέρη της Ευρώπης ε, αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Ε, έχουμε δει την μοτζαρέλα από την Ιταλία, ε, χείριο προϊόντα στην Ιρλανδία και προϊόντα βόλιο κρέατος από την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό που θέλουμε να δούμε και να τονίσουμε είναι ότι και πάλι απέτυχε να προστατεύσει τους καταναλωτές. Τι θα κάνει για να διορθωθεί η κατάσταση η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Δανέλης. Για ένα λεπτό κύριε επίτροπε δώδεκα χρόνια μετά το σκάνδαλο διοξινών στις βελγικές ζωοτροφές τώρα εντοπίστηκαν σε ζωοτροφές στη γερμανία χώρα με παράδοση στην πειθαρχία και τους αξιόπιστους θεσμούς. αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ελέγχων δεν είναι επαρκώς αυστηρό στοχευμένο διαφανές και αντικειμενικό και δεν συνοδεύεται από επαρκή αντικίνητρα και κυρώσεις. τα κενά αυτά πρέπει να καλυφθούν με σοβαρότητα και ευθύνη έναντι του καταναλωτή ιδιαίτερα σε μια εποχή που η οικονομική κρίση ευνοεί την εξέβρεση αθέμητων λύσεων για μείωση του κόστου παραγωγής δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι ιδιαίτερα σε αντίξωε οικονομικέ συνθήκε τα προβλήματα θα αυτορυθμίζονται στη βάση ενός συστήματος ηθικών αξιών και βέβαια οι καταναλωτές πρέπει να έχουν άμεση και πλήρη πληροφόρηση για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται η ευρωπαϊκή ένωση υπερηφανεύεται ότι έχει θεσπίσει αυστηρού όρου για τη διασφάλιση δημόσια υγεία τη προστασία του περιβάλλοντο τη ευζοία των ζώων. θα πρέπει όμω και να διασφαλίσει την απαρέγκλητη εφαρμογή του εάν δεν θέλει η πολιτική τη να περιοριστεί απλώ. Um. Ο χρόνο σα ε, τελείωσε. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται εδώ περί αμελίας. Εδώ υπάρχει ποινική ευθύνη. Οπότε εδώ πέρα χρειάζεται κάποιο είδου υποχρεωτική εντοκιοθεσία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην λέει μόνο τον τρόπο προέλευση, αλλά να υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε. Αλλιώ υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτού. Έχουμε και κάποιε μελέτε που αποδεικνύουν ότι ο καταναλωτή θέλει να ξοδεύει αν ε, ξέρει όμω τη διαδρομή του προϊόντο. Να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι. και τελικά δεν ε, βρήκε το τι συμβαίνει η εταιρεία ή συγγνώμη, η υπηρεσία για τι στροφές το βρήκαν οι ίδιες οι εταιρείες. Είναι σαφή η κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι για οτιδήποτε έχει σχέση με ζωικές στροφές και αφορά και του ανθρώπου. Και τώρα θα κάνουμε τη διαδικασία του Catch the Eye. Περίπου 40 συνάδελφοι μου ζητήσει το λόγο. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο γιατί βρισκόμαστε ελαφρώς πίσω στον όλο το χρονοδιάγραμμα άρα μίλησαν δύο από το ΕΛΚ και δύο από τους ε, ε, συντηρητικούς μεταρρυθμιστές για να μπορέσουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη ισορροπία και επίση να δούμε και τι θα γίνει με αυτού που έχουν ζητήσει το λόγο. Να δεν παρίστανται. Ο πρώτο ομιλητή τώρα θα είναι η κυρία Μακ Γκίνε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε στην Ιρλανδία. Πριν από δύο χρόνια, το 2008 Δεκέμβριο, υπήρχε πρόβλημα. Τι έκανε μέσα αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν η Κομισιόν για να αποφύγει τη σημερινή κρίση, συγκεκριμένη είναι η ερώτηση. Οι Εθνικέ αρχέ ε, διψάνε για κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά τις ε, ζωοτροφές. Να, να δώσετε και τις γραμμές, να φτιάξετε εργαστήρια. Δώστε τους αυτό που θέλουν. Κάτι άλλο τώρα. Θα πρέπει σίγουρα να εντοπιστούν τα προϊόντα υψηλού κινδύνου, οι διαδικασίες που έχουν υψηλό κίνδυνο και να ξέρουμε και πού βρίσκονται και ποιοι είναι η παραγωγή υψηλού κινδύνου. Και χρειάζεται 100% διαχωρισμός των προϊόντων που είναι να πάνε ε, σε ζώα και σε ζωοτροφές. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για, για, για μιλάμε για κάτι που έχει σχέση με τη, με, με, με τη ζωή μας, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα παίρνοντας με τη ζωή μας. Ε, καμιά φορά η εξοικονόμηση φέρνει φύρα. Ευχαριστώ. Πέρασε το ένα σας λεπτό. Κυρία Κάντμπαχ. Ένα λεπτό επίσης. Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύω στα, στις δηλιακές εικόνες των ευτυχών ε, πουλερικών ε, που χαμογελαστά πηγαίνουν ε, στη φάρμα. Όχι, γιατί ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Πλην όμω έχει μεγάλη σημασία να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόφιμα ασφαλή. Και γι' αυτό η κύρια μου, το κύριο μου αίτημα είναι αυστηρή έλεγχη και πιο, αυστηρή, πιο αυστηρές κυρώσεις. Βλέπουμε όμως δυστυχώ ότι δεν υπάρχει η γεωργική δομή που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσουμε και προς μια γεωργική μεταρρύθμιση διδασκόμενη από τα σκάνδαλα που βλέπουμε τώρα και να δώσουμε δομές μέσα στη γεωργική μας ε, δομή, μέσα στη γεωργική μας οικονομία η οποία θα εξασφαλίζει και την επιβίωση των γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και ασφαλή τρόφιμα. Και θα παρακαλέσω από το σκάνδαλο αυτό να αποκομίσουμε όλοι τα σωστά διδάγματα. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, κύριος Ασχούρθ, και ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε διάφορα περιστατικά όπως και αυτό εδώ και χρόνια και φανταζόμουν ότι μέχρι στιγμής η σημασία της ανιχνεσιμότητας και της εξασφάλισης ποιότητας θα είχε γίνει σαφώς κατανοητή και ότι θα υπήρχαν οι κατάλληλες δομές αλλά και οι κανονισμοί ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα. Αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρέ ανησυχίε. Καταρχήν, είναι ιδιαίτερα βλαβερό για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, βιομηχανία τροφίμων. Έπειτα, είναι πάντοτε οι αγρότε, οι, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι οι αθώοι ε, και οι οποίοι υποφέρουν από δυσανάλογες απώλειες, ζημιές λόγω τέτοιων ε, περιστατικών. Είμαι σχετικά ικανοποιημένο που οι γερμανικέ αρχέ και οι Κομισιόν έλαβαν λογική, ε, προχώρησαν μάλλον σε λογική και ταχαία δράση μόλι γνώρισαν, ανακάλυψαν το πρόβλημα. Ωστόσο, προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά ορισμένων τομέων της μεταπητικής βιομηχανίας, όπου σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερο όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και την σώρευση εξιών. Ευχαριστώ, έχει τελειώσει το ένα σας λεπτό, χρόνος ομιλίας σας. Και παρακαλώ τώρα τον κύριο Φερέιρα να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ανακάλυψη μολυσμένων προϊόντων από διοξίνε και η διάδοσή του μέσω διάφορων ε, καναλιών εμπορευματοποίηση αποτελούν μεγάλο ε, και πολύ σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ευθύνε, αλλά και ποιε είναι οι συνέπειε αυτού του γεγονότο και προχωρήσουμε σε ένα πιο βαθύ προβληματισμό όσον αφορά την αποτυχία ολόκληρου του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Έχουμε τι συνέπειε μια γεωργική πολιτική, η οποία είναι προσανατολισμένη μόνο στην αγορά, προωθεί πρότυπα εντατική παραγωγή, ε, ευνοεί την μεγάλη αγροβιομηχανία και εξαφανίζει την μεσαία και την οικογενειακή γεωργία και ευνοεί επίσης την ευρεία κατανάλωση όχι, ενώ δεν ευνοεί καθόλου την τοπική ε, κατανάλωση που εγγυάται πολύ πιο ασφαλή προϊόντα. Θέλουμε λοιπόν να επιβάλλουμε, να επιβληθεί μάλλον μια βαθιά αλλαγή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Σταραμπέλο Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς δικαιολογημένα να εκφράζει την ε, δυσφορία του για αυτές τις επανειλημμένες ε, κρίσεις που έχουν ταρανίσει άλλωστε και το Βέλγιο πριν από περίπου 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να έχουμε μέτρα πιο ε, αυστηρά ως προς τη λειτουργία του πλαισίου αλλά ως προς τις κυρώσεις γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια τυχαία ε, παράληψη. Έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερα εις βάρος της ζωής των άλλων. Και επίσης θα έπρεπε να δούμε και το ζήτημα της διακινδύνευσης. Και όπως είπε και η συνάδελφος το RABEX, δηλαδή το Rabbit Exchange, το σύστημα εκείνο το οποίο θα επιτρέπει, ε, εάν λειτουργήσει σωστά βέβαια, να ενημερώνονται τα κράτη το ένα από το άλλο, ε, για ορισμένους κινδύνους που φαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν λειτουργήσε ικανοποιητικά. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Γιάος, τελευταίος ομιλητής για τη δικασία του Κατστιάη. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η γερμανική ε, βιομηχανία τροφίμων έχει ένα ικανοποιητικό σύστημα αυτοελέγχου, το οποίο όμως δεν λειτουργεί όταν υπάρχει εγκληματική δράση, όταν έχει κανείς εγκληματική πρόθεση. Και ως εκ τούτου στην ε, ανάμιξη ε, βιομηχανικών λοιπόν μέσα σε ζωοτροφές έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να υπαχθεί σε οποιονδήποτε έλεγχο, θα διέφευγε από οποιονδήποτε έλεγχο δηλαδή. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι τακτικές περισσότερες ελεκτικές δραστηριότητες από το κράτος. Χρειάζεται επίσης να δημοσιεύονται υποχρεωτικά τα αποτελέσματα των ε, αναλύσεων σε ε, τρόφιμα και χρειάζεται για τους εγκληματίες αυτού που προβαίνουν σε αυτές τις εγκληματικέ πράξεις πιο αυστηρές κυρώσει, έτσι ώστε να σκέφτονται δύο φορέ πριν διαπράξουν το έγκλημα αυτό. Και κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι εκείνοι οι οποίοι περισσότερο υποφέρουν από αυτή την τελευταία κρίση είναι οι γεωργοί, εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στη θέση να διαθέσουν τα προϊόντα του, γιατί είναι αξιόλογα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο Επίτροπος Νταλή, τώρα εκ μέρους Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν συμμετέχω σε τέτοιες συζητήσεις δεν μπορώ παρά να προσέχω κυρίως τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν εις βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόλης της ύλης που μας κατηγορείτε ότι έχουμε γραφειοκρατία. Και λέτε ότι θα πρέπει να προβλέπουμε ελέγχους. Ο κλάδος όλοι γκρινιάζουν ότι εμείς δημιουργούμε γραφειοκρατία. Πάντως σε περιπτώσεις όπως η παρούσα διαπιστώνεται ότι οι έλεγχοι που υπάρχουν είναι πάρα πολύ αναγκαίοι. Χρειάζονται, είναι αναγκαίοι και θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηροί. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμόζονται. Και εγώ ίδιος είμαι καταναλωτής και δεν θέλω να βρίσκομαι σε κατάσταση όπως η παρούσα. Γιατί αισθάνομαι απειλή και χάνω την εμπιστοσύνη μου στα προϊόντα της αγοράς. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ολόκληρος εγκληματικός κλάδος που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων. Και όπως είπε ο τελευταίος αγορητής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όταν έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν οργανωθεί για να παραβιάζουν τον νόμο και δεν μπορεί να έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι στεγανό και υπάρχουν εγγυήσει ότι όλα λειτουργούν άριστα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μα για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε όσο γίνεται λιγότερα παραθυράκια στο σύστημα. Και έτσι οι εγκληματίε δεν μπορούν να ξεκλειστρήσουν. Εγώ ασχολούμαι με την νομοθεσία εδώ και 20 τόσα χρόνια. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι οι ρήτε που προβλέπονται, αλλά το να προσπαθεί κανεί και να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται. Καθώ επίσης και τα δίκτυα ασφαλείας τα οποία πρέπει να υπάρχουν ούτως ώστε να μην συμβαίνουν παραβιάσει. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να έχουμε σύστημα που δεν επιτρέπει σε αυτούς που επιδιώκουν την παραβίαση του νόμου να το κάνουν ατιμόρυτα. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται γνωρίζοντας το τι συμβαίνει. δουλεύει τώρα απ' Τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε, τη στιγμή που μάθαμε τι συμβαίνει, όλα πήγαν καλά. Θα πρέπει επίση να τελειοποιηθεί ο ισχυρό κανονισμό. Συμφωνώ. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνε. Μα είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι γραμμέ και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τέτοια στοιχεία δεν θα υπάρχουν στη διατροφική αλυσίδα. Και μακάρι να γίνουν όλοι σχετικοί έλεγχοι, ώστε να υπάρξει αποφυγή του κινδύνου. Επομένω, οι εταιρείε του κλάδου να μην καταγορούνται στο Μητρό των Εταιριών με απλή δήλωση, αλλά να προηγούνται τη έγκριση λειτουργίας τους έλεγχη. Πώς θα να καταδείξουμε ότι υπάρχουν οι, κατα... οι απαιτούμενοι έλεγχοι και είμαστε σε βέβαια επαφή με τις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία. Είμαι θα ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν τόσο ώστε να συγκρατηθεί αυτή η κατάσταση. Όσο γίνεται γρηγορότερα να αποκατασταθεί. Θα πρέπει να μάθουμε ακριβώ πώ έχει η κατάσταση των νεότερων δυνατών και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ο δε παραγωγό ο οποίος έχει παράσχει λανθασμένες πληροφορίες και ο οποίος έχει προμηθεύσει με ελαττωματικό προϊόν 900 εκμεταλλεύσεις ήδη είναι κατηγορούμενος και το έχει ασκηθεί πριν κυρίες βάρος του στη Γερμανία. Πάμε θα γίνει με τις εξαγωγές και τα αυγά. Που χρησιμοποιούν στον κλάδο των, ε, της μεταποίησης των τροφίμων. Ε, εδώ έχουμε ανάμειξη πολλών προϊόντων και προϊόντων που δεν ήταν γερμανικά. Και άρα το τελικό επίπεδο ιδιοξύνηση ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Τελευταίο σχόλιο τώρα. Συμφωνώ. Θα πρέπει να έχουμε αυστηρές κυρώσεις εναντίον όσων εκμεταλλεύονται το σύστημα. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το θεσπίσουμε μόνοι μας εμείς, ούτε να το επιβάλλουμε. Τα κράτη-μέλη οφείλουν εφαρμόσουν νομοθεσία στη χώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η κοινή συζήτηση για τη δασική νομοθεσία.